Das gilt auch für Sie, Herr Ναι, κύριε Φλέκενστάιν, και εσείς ήσυχος να είστε. Κυρίσω λοιπόν την άνοιξη της συνεδρίασης, έκτακτη συνεδρίασης, με θέμα πρόταση, δέσμη προτάσεων για την διεύρυνση και ρωτώ εάν υπάρχουν παρατηρήσεις στην ημερήσια διάταξη ούτε η Προεδρία έχει τίποτα, από πλευρά του Προεδρείου δηλαδή έχουμε τίποτα να παρατηρήσουμε για την ημερήσια διάταξη, το από εσά βλέπω. Επομένω, περνάμε στην ημερήσια, στο πρώτο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Φιούλε και παρακαλώ ε, ξεκινώντας να μου επιτρέψετε να τον ευχαριστήσω προσωπικώς για την ε, πενταετή αφοσίωση του στη δουλειά αυτή, στο έργο αυτό, σε συνθήκες δύσκολε με ριζικές αλλαγές, και αυτό το λέω έχοντας υπόψη την πολιτική γειτονία και βέβαια με το νέο χαρτοφυλάκιο το οποίο τώρα εκφράζεται ε, με τους όρους αυτούς και για την Ουκρανία και για την νότια γειτονία έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Δεν χρειάζεται να σας τις εκθέσω περισσότερο και βέβαια η διεύρυνση τελευταία με τη συμμετοχή της Κροατίας και οι προοπτικές των λοιπόν κρατών ήταν μεγάλες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν, σας συγχαίρω ταυτόχρονα και θα ήθελα ιδιαίτερος να σημειώσω ότι αποτελέσατε και ένα πολύ θετικό σήμα του πώς συνεργάζεται κανείς από την Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορίσατε ψηλά τον πύχη της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο. ως πρόεδρος της Επιτροπής μόνο περιστασιακά χρειάστηκε να εκδηλώσω διαφωνία μαζί σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό πάντα να συμφωνούμε. Πάντως διαπιστώνουμε ότι υπήρχε πνεύμα εμπιστοσύνη, κοινέ κατευθύνσεις, κοινή προσανατολισμοί και πνεύμα εξυπηρέτηση του συμφερόντος Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα από αυτό που έχουμε δει από ορισμένου, όπως είπατε, εκπρόσωποι Ο κύριος Φίλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Έλμαρ για τα καλά σου λόγια. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, βουλευτές, κυρίες και κύριοι, φίλοι της διεύρυνσης, αυτές τις μέρες στρέφω το βλέμμα πίσω προς άλλες ακροάσεις που είχα υποστεί ως υποψήφιος επίτροπος εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουν κλείσει περίπου πέντε χρόνια από τότε που ανέλαβα μια ισχυρή δέσμευση απέναντί σας για τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονία. Και χάρη στη δική σας στεναρή υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια μπόρεσα την δέσμευση αυτή να τη μετατρέψω σε δράσεις. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω την τελευταία πενταετία με τα πακέτα για τη διεύρυνση. Το 2010 ξεκινήσαμε τη δουλειά μας με εστίαση στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης. Το 2011 συνεχίσαμε με την έμφαση στην ενίσχυση της ε, δύναμης μεταλλαγής, μετατροπής που μπορούσε να φέρει η διεύρυνση. Αλλά βέβαια η δυσκολία ήταν να διατηρηθεί η ίδια έμφαση στις αρχές αυτές μακροπρόθεσμα και έτσι στηρίξαμε ιδιαίτερο στους τρεις πυλώνες κράτος δικαίου, οικονομική διακυβέρνηση και μεταρρύθμιση στις δημόσιες, στο δημόσιο φορές, στους δημόσιους φορείς. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το χτίσιμο του πρώτου πυλώνα, τη νέα προσέγγιση στο κράτος δικαίου και νέα στοιχεία αυτής της νέας προσέγγισης είναι ότι μια υποψήφια χώρα, μια χώρα που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του άρθρου 23 για τη δικαιοσύνη και του 24 για τη δικαιοσύνη 23 για τα ιστορικά και 24 για τη δικαιοσύνη και τις ελευθερίες έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Προεπραγματεύσεων επιμείναμε ιδιαίτερο σε ορόσημα, σε παρακολούθηση τήρησής τους και σε ρήτρε ισορροπίας. Το 2013 θεσπίσαμε ένα πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα από τους τρεις, την οικονομική διακυβέρνηση. Η προσέγγιση μας εμπνεόμενη από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο προτείνει από το επόμενο έτος καλύτερη καθοδήγηση, κυρίως για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σε θέματα φορολογικά και συμβατότητας και ιδιαιτέρως για εφέτος θα ήθελα να δώσω την έμφαση για τον τρίτο, στον τρίτο πυλώνα, μεταρρύθμιση των, του, κρατικών υπηρεσιών, του δημοσίου δηλαδή, ε, θεσμοί, υγιής διαχείριση, λογοδοσία των υπηρεσιών, που αποτελούν ε, κέντρο κάθε ορθώς λειτουργώντος κράτους. Έτσι λοιπόν οι χώρες ενθαρρύνονται να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς. Οι τρεις πυλώνες της διαδικασίας της διεύρυνσης που σας περιέγραψα ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Πρόοδος δηλαδή στους τομείς αυτούς θα αποτελέσει και κλειδί για την αξιολόγηση του πότε μπορεί να είναι έτοιμη για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, αυτό ήταν το βασικό πλαίσιο. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω σε άλλα σημαντικά θέματα που θα δείτε και στο έγγραφο στρατηγικής που εκδόθηκε φέτος. Καταρχάς λοιπόν έχουμε την σημασία της, της, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθερία έκφρασης, προστασία ευάλωτων ομάδων. Δεύτερον, υπογραμμίσουμε την σημασία της περιφερειακής συνεργασίας η οποία επιτρέπει στους εταίρους μας να προωθήσουν τις ε, πραγματικές προτεραιότητες με επενδύσεις και συνεταιρικές ε, σχέσεις μέσα στην περιφέρειά τους, αλλά και από την περιφέρειά τους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες θετικές εξελίξεις του περασμένου έτους στον τομέα αυτό έχουν να κάνουν με την συμπερίληψη όλο και περισσότερο του κοσμοπεδίου σε περιφερειακά κέντρα συζητήσεων, το ρόλο των δυστικών ε, Βαλκανίων στην ενισχυμένη συνεργασία στην διαδικασία σύνδεσης, ε, και τη Σύνοδο του Βερολίνου του Αυγούστου η οποία επικεντρώθηκε στην περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία και θα ήθελα να σημειώσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι προβλέπονται και άλλες ε, τέτοιες σύνοδοι με ε, οικοδεσπότη αυτή φορά την Αυστρία. Τρίτον, σε όλη μου την θητεία ιδιαίτερη έμφαση και σημασία απέδωσα στην ελευθερία έκφρασης, όπως άλλωστε και το Κοινοβούλιο το 2011 και το 2013, τη δέσμευση αυτή την υπογραμμίσαμε, την εκφράσαμε, ε, οργανώνοντας τις διασκέψεις «Μίλα δυνατά, ύψος τη φωνή σου». Τώρα όμως θα πρέπει και να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για, τους, ε, για τις προκλήσεις που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ως προς την ελευθερία έκφρασης, τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και στην Τουρκία. Τέταρτον, υπογραμμίζουμε τη σημασία επικοδομητικού και αηφόρου διαλόγου σε όλο το πολιτικό φάσμα στις χώρες που θέλουν να ανταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια σειρά ε, διαλόγων διαρθρωμένων σε υψηλό επίπεδο που γεννούν περισσότερες ευκαιρίες για τις χώρες ώστε αυτές να αναπτύξουν μεταρρυθμίσεις και βέβαια από πλευράς μας εμείς θα τους προσφέρουμε την αρρωγή μας. Πάντως, διαπιστώνεται μία τάση όπου βλέπουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τα κοινοβούλια δεν συμμετέχουν στην διαδικασία αναμόρφωσης των δημοκρατικών θεσμών. Μποϊκότ δηλαδή. Και μπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονη ε, διαμαρτυρία αυτό, το μποϊκότ, σαφή διαμαρτυρία, σαφής διαμαρτυρία, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων. Η μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών είναι ευθύνη και των δύο πλευρών. Κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Και πρέπει οι κυβερνήσει αυτές να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα για την αντιπολίτευση πλήρω να εκτελέσει το δικό της μέρος του δημοκρατικού ελέγχου, της λειτουργία του δημοκρατικού ελέγχου, όπως είναι και ε, καθήκον των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν με τρόπο επικοδομητικό σε αυτέ τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Πέμπτον. Στο νέο μέσον προενταξιακής ενίσχυσης, το είπα έχουμε αξιοποιήσει πολύ περισσότερο την υποστήριξη τη δημοσιονομική με μια τομεακή προσέγγιση και θα αξιολογήσουμε τις καλές επιδόσεις με βάση την ανταμοιβή για τις επιδόσεις, εάν θέλετε να το πούμε έτσι. Τώρα πριν περάσω στις επιμέρους ε, χώρες, χώρες ήθελα να συμμεριστώ μια ιδέα που με απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Και όσον αφορά τις πρόσφατες ε, συζητήσεις για το τι θα είναι μια λογική ε, αρχή, ένα λογική όρη του παιχνιδιού για τη διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας θυμίσω λοιπόν αυτά που λέγαμε τον πρώτο χρόνο της εντολής μου, όπου λέγαμε ότι άπαξ και η χώρα υποψήφια, η ενδιαφερόμενη για τη διεύρυνση προχωρήσει στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και εμείς προχωρούμε στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών προοπτικών. Έτσι η αξιοπιστία είναι αμφίδρομη και δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων στα ανατολικά της Υπήρου μας, είναι όλο και πιο ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμήσει αυτή την αρχή. Κυρίες και κύριοι, περνάω τώρα στις ε, χώρες επιμέρους. Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει ακόμα 10 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων συμπεριλαμβανομένων και των υπαριθμών 23 και 24. Η υλοποίηση του κράτους δικαίου ε, και οι σχετικές μεταρρυθμίσεις έχει ξεκινήσει με την, υλοποίηση, με την εισαγωγή μάλλον νομοθεσίας και μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δικαιοσύνης. Οι προθεσμίες όμως δεν τηρούνται επαρκώς σε διάφορους τομείς και τώρα το Μαυροβούνιο πρέπει να προχωρήσει σε κατεπίγουσα δράση, ανάληψη δράσεως για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα κράτος δικαίου και συναφή ζητήματα και ανάγκη για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης με ένα σταθερό βήμα στις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου που θα καταστεί κέρια σημασία για την αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχει ικανοποιητικός ρυθμός στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη η νομοθεσία για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων θα έχει πολύ μεγάλη σημασία εφόσον μεταρρυθμιστεί ικανοποιητικά δηλαδή και η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου έτσι ώστε να, μπει στην, ε, ε, να ρυθμιστούν τα ζητήματα αυτά της δημοκρατικής διαδικασίας. Έχουμε μια μεταρρύθμιση που εχθές μόλις, ύστερα από πολλαπλές ε, απόπειρε ενέκρινε το Κοινοβούλιο και έτσι μπορούν πλέον οι θεσμοί να καταγράψουν θετικές ε, θετικά αποτελέσματα ως προς την δίωξη της διαφθοράς και των σχετικών εγκλημάτων. Σερβία, όπου έχουμε μια σημαντική αλλαγή τα τελευταία χρόνια με αναγνώριση των προόδων που έχει επιτύχει η Σερβία τόσο στην, στο θεματολόγιο για τη μεταρρύθμιση όσο και ως προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με το κοσμοπέδιο. Ως ε, χώρα διαπραγματευόμενη την ένταξη. Η Σερβία έχει και ευθύνε αλλά και νέε ευκαιρίε να δράξει. Η Σερβία έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο δέσμευση και επαγγελματικότητα και, και στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων με την διαδικασία του screening, τη επαλήθευση νομοθεσία που συνεχίζεται απρόσκοπτα. Τώρα πρέπει να συνεχίσει να προχωρεί στις, ε, στην υλοποίηση μάλλον των προτεραιοτήτων για, για τις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο κράτο δικαίου, τη δημόσια διοίκηση αλλά και την οικονομική διακυβέρνηση και είναι πολύ σημαντικό η Σερβία να συνεχίσει τι δεσμεύσει τη ω προ την περιφερειακή συνεργασία και την εξομάλυνση των σχέσεων με το Πρέπει να δοθεί νέα όθηση για να αντιμετωπιστούν κέρια σημασία σε κρεμή ζητήματα και να ανοίξει μια νέα, να ξεκινήσει μια νέα φάση στην διαδικασία της εξομάλυνσης. Αυτό έχει κέρια σημασία για τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουν λοιπόν απρόσκοπτα αυτές τις διαδικασίες. Με αυτές, σε αυτές τις προσπάθειες η Σερβία μπορεί να στηρίζεται στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται μετά τις πολύ σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την Σερβία το Μάιο δείχνοντας ότι είναι διατεθειμένη και αποφασισμένη να σταθεί στο πλευρό της Σερβίας σε κάθε πρόβλημα όσον αφορά την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η διαδικασία Ευρωπαϊκή, ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει σε αδιέξοδο. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η οπισθοδρόμηση σε κέριους τομείς μεταρρυθμίσεων που ε, εμφανίζεται στο τελευταίο έτος. Παραμένει ουσιώδου σημασία να αναλυφθούν καθοριστικά βήματα για την επίλυση του προβλήματος του ονόματος με την Ελλάδα του ζητήματο του ονόματος από την Ελλάδα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η διαδικασία υπό τα Ηνωμένα Έθνη για την επίλυση του προβλήματος αυτού, του ζητήματος αυτού, ε, έχει ξεκινήσει εδώ και 19 χρόνια. Διατυπώνονται συστάσεις για την έναρξη των ε, διαδικασιών διαπραγματεύσεων. Πρέπει η χώρα να συνεχίσει για να ευθυγραμμιστεί στις προϋποθέσεις, να πληρεί τις απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις, Ταυτόχρονα όμως τα Σκόπια θα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση εάν επιθυμεί να εξασφαλίσει την θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον. Αποφασιστική δράση απαιτείται για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες, όλο και αυξανόμενες ανησυχίες για την εντυνόμενη πολιτικοποίηση και ε, τα προβλήματα τα σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ελευθερία της έκφρασης τα κομματικά συμφέροντα επικρατούν των εθνικών συμφερόντων από ό,τι φαίνεται. Πρέπει ο πολιτικός διάλογος λοιπόν να διεξάγεται κατά κύριο λόγο στο Κοινοβούλιο και να συνεχίσει να ε, εξυπηρετεί τον κύριο αυτόν στόχο του δημοκρατικού διαλόγου. Συνεχίζονται, ελπίζουμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε τη χώρα στη συνέχιση των προσπαθειών της για έναν ε, πλήρη διάλογο για την ένταξη που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, μεταρρύθμιση. Η Αλβανία έχει εξασφαλίσει το καθεστώς του υποψηφίου κράτους στον Ιόνιο. Η κυβέρνηση επιδεικνύει βούληση για ένταξη και υλοποίηση των ε, μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ένταξη. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών με εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις αστυνομικές αρχές αποδεικνύει τη βούληση της χώρας να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Μας ανησυχεί όσο ωστόσο η επιδείνωση του πολιτικού κλίματος και το μποϊκότ της αντιπολίτευσης από, τα από το κοινοβουλευτικό έργο. Θα πρέπει η κυβέρνηση να επιτρέψει στην αντιπολίτευση να εκτελέσει πλήρως τους, ε, τις λειτουργίες του δημοκρατικού ελέγχου το καθεστώς του υποψηφίου κράτους ενέχει περισσότερες ελπίδες και μπορεί να αποτελέσει και κίνητρο για την επιτευξή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση τώρα θα πρέπει να αποδείξει ότι διατηρεί τις δεσμεύσεις της για μεταρρύθμιση και για ουσιαστικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, καθώς και πώς κάνει ό,τι μπορεί ώστε να επικρατήσουν συνθήκες διαφάνειας και ανοιχτού πολιτικού κλίματος. Η Βοσνία Σεγοβίνια το τελευταίο χρόνο έχει κάνει πολύ περιορισμένη πρόοδο, δεν υπάρχει πολιτική κινητικότητα και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με, τη βούληση και τη θέληση των πολιτών της Βοσνίας Σεγοβίνης να δουν μια πρόοδο στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις, γενικές, ε, τις επικείμενες γενικές εκλογές θα είναι πολύ σημαντικό να σχηματιστούν ταχύτατα όλα τα όργανα σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης έτσι ώστε η χώρα ταχύτατα να βρει τρόπους αποτελεσματικού συντονισμού και αντιμετώπισης των κατεπηγουσών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και βέβαια υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης. Μόνο με σημαντική πολιτική κινητικότητα και όθηση μπορεί η Βοσνία Ερσεγοβίνη να ξεπεράσει την ε, στασιμότητα στη διαδικασία για την ε, ένταξη. Η Συμφωνία Σύνδεσης ε, και Συνεργασίας του Ιουλίου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου, το Κωσυφοπέδιο πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα του ρυθμού, δεν έχει περιθώριο να καθυστερήσει, γιατί τα διακυβευόμενα είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά. Έτσι λοιπόν, πρέπει ταχύτατα να αναλάβει δράση ο νόμοθέτης, γιατί αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα αποτελεί δρόμο σε σχέση με τι μεταρρυθμίσει. Το αδιέξοδο μετά τι εκλογέ, πρέπει να αντιμετωπιστεί και να θεσπιστεί ταχύτατα κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να εκπληρώσει τις ε, να υλοποιήσει τις πρόπτικες της, ε, του κοσμοπεδίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσει ένα διάλογο ανοιχτό και ε, χωρίς αποκλεισμούς για τη μεταρρύθμιση και, στο, και την υλοποίηση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και την υλοποίηση της του θεματολογίου για την οικονομική διακυβέρνηση. Όπω είπα και νωρίτερα, νέο, νέα όθηση θα πρέπει να χορηγηθεί και στον διάλογο, πρέπει να δοθεί στον διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κουσποπεδίου για να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ακόμα ζητήματα και να προχωρήσουν οι δύο χώρες σε μια εξομάλυνση των σχέσεών του για την Τουρκία. Έχουν υλοποιηθεί αρκετά θετικά βήματα το τελευταίο χρόνο, θετικά και φιλόδοξα βήματα για την αντιμετώπιση του κουρδικού προβλήματος. Το 2013 είχαμε το πακέτο για τον εκδημοκρατισμό. Θέλω επίσης να σημειώσω την θέση σε ε, εφαρμογή μιας συμφωνίας ε, επαναπροώθησης, επανεισδοχής, το θέμα των θεωρήσεων των διαβατηρίων και το, την υποδοχή από πλευρά της Τουρκία, έως και ενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Συρία. Τους τελευταίους μήνες όμως σημειώνονται εξελίξεις οι οποίες ε, προξενούν ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προτάσεις για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, όπως τροποποίηση στο δίκαιο το σχετικό με το διαδίκτυο, οι γενικευμένες απαγορεύσεις του Twitter και άλλων ε, κοινωνικών δικτύων μας ανησυχούν ιδιαίτερως. Ιδιαίτερα δε καθώς χρησιμοποιούνται ειδικά ποινικά δικαστήρια και ο αντιτρομοκρατικός νόμος για τον ε, περιορισμό, για την περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης, ρυθμιστικές αρχές ακόμη βλέπουμε που ότι ενώ έχουν συσταθεί δεν έχουν ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα που αποτελούν επίσης λέξεις κλειδιά για την δικαιοσύνη και πρέπει να ενισχυθούν. Η παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων της Τουρκίας από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας θα πρέπει να αποφεύγεται χωρίς ε, μεταβατικές ε, ρυθμίσεις γίνονται μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές ε, στη λειτουργία των δικαστηρίων που θα έχουν σαφέστατες συνέπειες στην πρόσκοπτη λειτουργία τους. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν μετακινήσεις και απολύσεις αξιωματούχων της αστυνομίας, δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών αυτών. Τούτου λεχθέντος, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναπόφευκτα ε, κοινό και το μέλλον. Είναι στρατηγικό εταίρος Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, όχι μόνο, αλλά πάνω απ' όλα για τι ε, οικονομικές και εμπορικές του σχέσεις, η, οικονομική, η περαιτέρω συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία έχει οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη να παραμείνουν ο κύριος μοχλός και η κινητήρια μηχανή για τις σχέσεις μας και γι' αυτό επαναλαμβάνω τη σύστασή μου να προχωρήσουμε με το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 που θα εξασφαλίσουν για την Τουρκία ένα σαφή οδικό χάρτη, ένα φύλλο πορείας για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στηριζόμενες στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Από την άλλη όμως θα πρέπει η Τουρκία να αποδείξει ότι προχωρεί με τρόπο συνεχή και σταθερό στις μεταρρυθμίσεις και ότι είναι σε θέση να τιμήσει τις πρόσφατα ανανεωμένες ε, δεσμεύσεις της για πρόοδο στη δημοκρατική μεταρρύθμιση. Για το θέμα της Κύπρου. Επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω και πάνω απ' όλα έχοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στην και γύρω από την Κύπρο. Ότι συνεχίζουμε την υποστήριξη των ε, γενικών συνομιλιών μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και της, ε, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Στις 11 Φεβρουαρίου είχαμε μια κοινή δήλωση με τον Άσπερ Μπαθ Άιντεν εκπρόσωπο απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το ζήτημα της ε, προώθησης των διαρθρωμένων συνομιλιών που αποτελούν μια θετική εξέλιξη. Μια συμφωνία λοιπόν για μια δίκαιη, βιώσιμη λύση και σταθερή λύση θα ενισχύσει σταθερότητα στην περιοχή, αλλά βέβαια θα αποτελέσει και σημαντικό κίνητρο και ε, σημείο όθηση για την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα θα ανοίξει και θα διευρύνει πολλέ επιλογέ ε, και δυνατότητε για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και θα προωθήσει κατά τον πιο ε, πλεονεκτικό τρόπο τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων. Η ελπίδα μου λοιπόν είναι πως θα αναλυφθούν επικοδομητικά βήματα ώστε να αποκατασταθεί και πάλι μια θετική ατμόσφαιρα γύρω από το θέμα των, ε, της ρύθμισης της επίλυσης του Κυπριακού. Ας περάσουμε τώρα από τις ε, χώρες ε, στους πολιτικούς. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου προς τους νέους συγητές ε, και να εκφράσω την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου σε όσους όλοι ήταν από την αρχή υπέρμαχοι και μεγάλοι φίλοι της διεύρυνσης και του αρμόδιου ε, επιτρόπου. Ο κύριος Κούκαν, που για πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ήταν επικεφαλής της και ήταν ανέκαθεν ε, πολύ διαλλακτικός και προσπαθούσε ανέκαθεν να κατευνάσει τα πνεύματα και στις πιο σφοδρές ε, συζητήσεις. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ, που ήταν ταυτόχρονα και υποστηρητικός αλλά και επικριτικός ε, απέναντι στη χώρα για την οποία είχε την, την έκθεση. Η κυρία Λούνατσεκ με το πάθος της και την αποφασιστικότητά της μας κράτησε όλους στην ατζέντα για το κοσυφοπέδιο. Τσάρλ Στάνοκ κάπου τον αφήσω το μάτι μου. Ένθερμος υποστηρικτής των συμφερόντων του Μαυροβουνίου και επίσης ε, απαιτούσε μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Πρέντα που ε, ήταν εισηγητής για μια χώρα που τελικά ε, ανέστηλε την, την το αίτημα της ένταξής της. Δεν ήταν εύκολο το έργο του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους φίλους της διεύρυνσης, που δεν είναι πια μέλη της Επιτροπής, Ντόρι Πάκρη, Όμεν Ρόιτεν, Φόλτον, Γιάλκο Κάτσεκ, Ρόουτσεκ, Νίκολα Βουλιάνιτς, Χάνεξ Σβόμποντα, Γιώργο Χατζημαρκάκης, Φραντσίσκα Χέρβεν, Εμινέ Μποσκούρτ, Μαρία Κορνέλισεν και δεν είναι εξαντλητικός ο κατάλογος. Και τέλος, αλλά ε, πολύ, σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έλμαρ Μπρόκ, τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο και σταματάω εδώ. Ήρθε κύριε πρόεδρε, κύριε και κύριοι η ώρα για την τελευταία μου ομιλία περί διεύρυνσης. Είπα ότι πριν από πέντε χρόνια ε, θέσαμε ως στόχο να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της ε, πολιτικής διεύρυνσης και τις ε, δυνατότητες μεταμόρφωσης που είχε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Έκτοτε αναζωογονήσαμε τη διεύρυνση και εκεί που θεωρούνταν μια τεχνική διαδικασία έλαβε μια τελείως διαφορετική ε, εικόνα και κρίθηκε ως κορυφαίο μέσο εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την τελευταία πενταετία η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά. Έχουμε μεγαλύτερη μεγαλύτερο ανταγωνισμό εκτός των σύνορων μας και χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις ε, στη, γειτονία μας. Και η διεύρύνση είναι ο καλύτερος χώρος για να το πετύχουμε. Η υποχωρητικότητα, η παρέτηση δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Και θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη και να προσφέρω την στήριξή μου και τη βοήθειά μου στον διάδοχό μου. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σας. Σε ευχαριστώ, Στέφαν. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στους εισηγητές και κατόπιν στους εκπροσώπους των ομάδων. Κριστιαν Πρέντο, εισηγητής για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι η τελευταία φορά που έχουμε την τύχη να σας έχουμε εδώ για την παρουσίαση του πακέτου διεύρυνσης. Θα ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σε ευχαριστήσω θερμά για όλες σας τις προσπάθειες τις τελευταίες πενταετίες προκειμένου να προωθήσετε τη διαδικασία διεύρυνσης. Τα τελευταία αυτά χρόνια είχαμε πολύ στενή συνεργασία. Δεν χάσατε καμία ευκαιρία για διάλογο με τους ευρωβουλευτές. Και φέτος η διαδικασία αξιολόγησης της πολιτικής διεύρυνσης έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί κάνουμε έναν απολογισμό της τελευταίας πενταετίας και προσδιορίζουμε τους βασικούς άξονες και της μελλοντικής μας πολιτικής. Και ο διάδοχός σας ε, θα πάρει επάξια τη σκήτα. Άλλη θα είναι καλός επίτροπος ο κύριος Χάν, θα συνεχίσει το έργο σας και το επιβεβαίωσε και στην ακρόαση που είχε στην Επιτροπή μας. Θέλει και ο κύριος Χάν να προβάλλει περισσότερο τα οικονομικά πλεονεκτήματα μιας μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη, τους λαούς στο χώρο της διεύρυνσης. Και αυτό το θέμα σας είναι και σας ιδιαίτερα προσφυλές. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές σκέψεις και να υποβάλω και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία της διεύρυνσης αυτή. Έχουμε μια δοκιμασμένη πια μεθοδολογία, εύρυθμη, που λειτουργεί σωστά και δεν πρόκειται να επιβάλλουμε κάποιες ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται όμως κάποιες βελτιώσεις. Να τονίσουμε περισσότερο τα απτά και ορατά αποτελέσματα που είχαμε στη διαδικασία της διεύρυνσης. Ποια είναι τα benchmarks, η συγκριτική κανόνες ή τα σημεία αναφοράς, τα ορόσημα για την έναρξη κάθε κεφαλαίου το διαπραγματεύσεων για κάθε κεφάλαιο και για την καταμέτρηση ή την αξιολόγηση των της προόδου του... της κάθε υποψήφιας χώρας. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία πιο ορατή και για τις υποψήφιες χώρες αλλά και το ευρωπαϊκό κοινό. Και ξεχάσαμε και εκτός από την ε, εμπέδωση, την αιρεσιμότητα και την επικοινωνία θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην επικοινωνία, να εξηγήσουμε δηλαδή τι σημαίνει κάθε στάδιο της διαδικασίας και για τις ε, υποψήφιες χώρες αλλά και για τις χώρες μέλη, ώστε να έχουμε ταυτόχρονη κινητοποίηση και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στεφθεί με επιτυχία η διεύρυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της διαδικασίας. Φυσικά δεν έχουμε ε, αντίστοιχη πρόοδο σε όλες τις χώρες. Είχαμε έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Σερβία, δόθηκε το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Αλβανία, είχαμε πρόοδο και φυσικά ε, επαναλαμβάνουμε ακούραστα ότι η διαδικασία αυτή ε, στηρίζεται σε επιδόσεις της κάθε υποψήφιας χώρας. Δεν θα πρέπει όμως ε, η πρόοδος να διακυβευτεί από κάποιες πολιτικές εξέλιξεις, γιατί η πολιτική πόλωση και η έλλειψη πολιτικού διαλόγου εξακολουθούν να είναι δεινά προβλήματα σε ορισμένες χώρες που έχουν ενταξιακές βλέψεις. Ε, θα σα θέσω ερώτηση για την Ισλανδία όπω σα έχω συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη που θα είναι η χώρα για την οποία θα κάνω έκθεση. Η ιστορία τη Ισλανδία δείχνει ακριβώς και η περίπτωση της Ισλανδίας δείχνει πόσο σοβαρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δέσμευση των υποψηφίων χωρών υπέρ της διαδικασίας ένταξης. Σε ό,τι αφορά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, είναι η δεύτερη συνέχεια χρονιά που διαπιστώνουμε πολύ περιορισμένη πρόοδο στα πολιτικά κριτήρια. Η θέση ισχύ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει καθυστερήσει. Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση είναι ανησυχητική και αυτό έχει φανεί και από τις ε, ε, διαδηλώσει στις αρχές του έτους. Οι φετινές πλημμύρες περιέπλεξαν την κατάσταση. Και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είχαμε σημαντικές ε, εντυπωσιακέ ε, μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων θεσμών. Και η οικονομική και πολιτική κατάσταση είχε αρνητικά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ενός μηχανισμού συντονισμού εν ώψη της ένταξης. Ξέρω ότι αφιερώσατε πολύ χρόνο και ενέργεια στο θέμα αυτό. Αλλά πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να βγει από το αδιέξοδο και να δημιουργήσει μια αξιόπιστη υποψηφιότητα για ένταξη. Νομίζω ότι μετά από μια πενταετία έχετε πολύ σημαντικά πράγματα να μας πείτε. Και χαίρομαι για την έκκληση που απευθύνατε ε, στην ένδειξη ελληνική μας προς την πολιτική τάξη της ε, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης εν ώψη και των ε, επικείμενων εκλογών, βουλευτικών εκλογών. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από, τις, ε, από τα πολιτικά και εθνοτικά χάσματα για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Βοσνία Ριζεγοβίνη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω για το συμφέρον της Βοσνίας ότι ο κύριος Μπρέντα θα είναι επιτυχής όπως και στην έκθεση για την Ισλανδία. Μα δεν φταίω εγώ κύριε Πρόεδρε. Μην υπερβάλλουμε το ρόλο του εισηγητή. Δεν έφταιγα εγώ. Και αυτό σωστό. Παρακαλώ τους αδέρφους όμως να είναι πιο σύντομοι τώρα. Ω συντονιστή εκ μέρου τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, παρακαλώ να αναλάβετε το λόγο ε, για την έκθεση που έχετε ο καθένα και παρακαλώ τον κύριο Φλέκενστάιν τώρα για την, για την Αλβανία να λάβει το λόγο. Κύριε Φίλε, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Βεβαίως θα υποστηρίξουμε τον διάδοχό σας ακριβώς όπως και εσάς, εφόσον δουλεύει τόσο καλά όσο και εσείς. Και αν όχι, θα πρέπει να κατευθύνεται και να προσανατολίζεται με βάση αυτά τα οποία καταγράφηκαν σε αυτά που μας είπε στην ακρόαση, όχι διεύρυνση και σφαλμένα μηνύματα, αυτά πρέπει να είναι η κατευθύνση Και επίσης επισημάνατε ότι η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο. Ιδιαίτερα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι σαφείς οι πρόοδοι και ορατές. Με το καθεστώς όμως του υποψηφίου κράτους η κυβέρνηση λαμβάνει, αναλαμβάνει νέες υποχρεώσεις, όπως και η αντιπολίτευση. Και θα πρέπει να παραμελήσουμε εδώ να επισημάνουμε στην Επιτροπή μας πόσο σημαντικό είναι να γίνει μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης να προχωρήσει ο αγώνας κατά της ε, διαφθοράς και πιο εντατικά και βέβαια να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδιαίτερος και σε πρώτη γραμμή των διακρίσεων εις βάρος των μειονοτήτων. Και σε αυτό το, με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει εμείς από πλευρά μας για να προσφέρουμε τη βοήθεια στους Αλβανούς φίλους που χρειάζονται. Αυτό ισχύει για την αντιπολίτευση όπως και για την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Τάνοκ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών τον Επίτροπο. Στέφεν, πράγματι έχεις δημιουργήσει μια χρήσιμη κληρονομιά για τον διάδοχό σου. Εύχομαι ε, λοιπόν καλή τύχη στις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα αναλάβεις στη ζωή σου. Ήμουν εισηγητής ε, εδώ και πέντε χρόνια για το Μαυροβούνιο και νομίζω ότι θα συνεχίσω και κάποια στιγμή δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει βέβαια με το δημοψήφισμα το 2017 αλλά ελπίζω να είμαι εδώ για να δω την πρόοδο στο Μαυροβούνιο. Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα πράγματα από το προηγούμενο κοινοβούλιο μέχρι σήμερα παραμένει στην ίδια κατηγορία του λεγόμενου το μικρό είναι όμορφο, σταθερή πολιτική σκηνή, καλά πηγαίνει η οικονομία και ο τουρισμός. Είναι μια εύκολη έκθεση που πρέπει να συντάξει κανείς εξ ονόματος της Επιτροπής μου και του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δεχτούμε, ιδιαίτερα μετά από τις τελευταίες ευρωεκλογές, ε, και τις αλλαγές που έγιναν στη σύνθεση του Κοινοβουλίου μας ότι υπάρχει η λεγόμενη κόποση της ε, ε, διεύρυνσης στο εκλογικό σώμα και γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε και τους εκλογείς μας γιατί η διεύρυνση είναι σημαντική για αυτές τις χώρες γιατί είναι κάτι το οποίο θα προσδέσει την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων στην σταθερότητα και την ασφάλεια στο μέλλον. Στην περίπτωση του Μαυροβουνίου χαίρομαι γιατί 12 από τα 35 κεφάλαια έχουν ανοίξει, δύο έχουν ήδη κλείσει. Η πρώιμη έναρξη του 23 και του 24 για τη δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις ήταν κάτι το πάρα πολύ θετικό γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και η έλλειψη της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος είναι μόνιμο πρόβλημα στην περιοχή. Η Βουλή του Μαυροβουνίου κατάφερε τελικά να εγκρίνει και τον διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τις ε, πιθανολογούμενες εκλογικές ε, αριθμίες. Λοιπόν, ελπίζω ε, να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και προσωπικά Στέφεν καλή τύχη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Φίλε για την παρουσίαση και το πεντατέστο έργο. Είμαι καινούριο Ευρωβουλευτής, αλλά γνωρίζω και το όνομά σας και το έργο σας. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από την ικανότητά σας ε, να δημιουργήσετε τόσο ευρεία συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της διεύρυνσης και ελπίζω και ο διάδοχός σας να συνεχίσει αυτή την πορεία. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πολιτικής μου ομάδας των Πρασίνων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τακτικές σας ε, ε, παρουσίες ε, στις συνεδριάσεις μας και την ε, άμεση και ειλικρινή επικοινωνία που είχαμε και τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει τις επαφές μας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ευχή της ομάδας μας μια γενική ευθύ για τη διαδικασία διεύρυνσης και όταν μια υποψήφια χώρα είναι έτοιμη και πρόθυμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρεί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουμε θεσπίσει για τις υποψήφιες χώρες, τότε ένα, μια απλή δήλωση στην, σε μια εκλογική εκστρατεία να μην εμποδίζει αυτή τη χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικώ είμαστε υπέρ τη διαδικασία διεύρυνση και ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια. Αντικαθιστώ εδώ την κυρία Τσέκ για την έκθεση του Κωσυφοπεδίου και θα ήθελα να σας μεταφέρω και τις δικές της ευχές και χαιρετισμού και να σας πω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι παρά την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει γίνει και σε επίπεδο κυβέρνηση ε, και σε επίπεδο κράτος δικαίου και εφαρμογή του δικαίου και χεγγύων κράτους δικαίου, πολύ δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Γιατί η, τα σώματα επιβολής του νόμου και η, δικαιοσύνη του κοσυφοπεδίου έχουν πολλές ε, αδυναμίες. Είχαμε ε, δεν είχαμε σταθερή ε, θέση του Κωσυφοπεδίου για τη συνεργασία ε, κάποιων δικαστών με το Συνταγματικό Δικαστήριο και ελπίζω να βοηθήσουμε την ενίσχυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στο Κωσυφοπέδιο. Επίσης, η μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τη Γιούλεξ στις τοπικές αρχές, που θα ολοκληρωθεί μετά από μια διετία. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή αναμένεται και νέα παράταση της αποστολής της Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner, for presenting the enlargement package. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μας παρουσιάσετε το πακέτο της διεύρυνσης. Θα είμαι ο νέος εισηγητής της έκθεσης ε, για τη Σερβία που συστηματικά πραγματοποιεί πρόοδο στην πρωταξιακή της διαδικασία. Έχει ξεκινήσει, μπήκε στις ράγες η διαδικασία αυτή και είναι σαφές ότι η Σερβία έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε όμως ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά περίπλοκα κεφάλαια και η Σερβία στο εγγύς μέλλον θα αντιμετωπίσει κυρίως ε, ε, δύο προκλήσεις, την εξομάλυση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο και το κράτος δικαίου. Η Συμφωνία των Βρυξελών ε, τον Απρίλιο ε, ήταν ε, ορόσημο στην εξομάλυση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας. Θα πρέπει όμως να συνεχίσει η Σερβία τις δεσμεύσεις και την υλοποίησή τους για να εφαρμοστούν ε, οι συμφωνίες και να ενισχυθεί ο διάλογος. Βέβαια, η έλλειψη κυβέρνηση στην Πρίστινα δεν διευκολύνει τη διαδικασία αυτή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τις Σερβικέ αρχέ ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει στο κράτος δικαίου, γιατί μια επαγγελματική ε, και ανεξάρτητη δικαστική εξουσία θα διαδραματίσει κύριο ρόλο στην πάταξη του εγκλήματος και τη διαφθορά. Θα πρέπει να συνεχίσει πέραν των μεταρρυθμίσεων του κράτου δικαίου και κάποιε οικονομικέ μεταρρυθμίσει, όπω την δημοσιονομική εξυγίαση και την αναδιάρθρωση ή ιδιωτικοποίηση κάποιων κρατικών ε, εταιριών. Θα πρέπει να τηρήσει λοιπόν τις υποχρεώσεις της Σερβία και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παραμένει σταθερά υπέρ της ε, διαδικασίας διεύρυνσης. Και στη διάρκεια των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αμέριστα τη Σερβία ε, με τα κονδύλια του μέσου προενταξιακής αρρωγής. Είμαστε ο σημαντικότερος δωρητής και σημαντικός εμπορικός εταίρος και θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία να αντιμετωπίσει ε, τι ζημίε από τις ε, καταστροφικέ πλημμύρε του Μαΐου. Σα ευχαριστώ. Αγαπητέ Επίτροπε, είμαι η συγγήτρια του νέου πλέον ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε η κυρία Ομεν στο παρελθόν να υπογραμμίσω επίσης και τις θαραλές θέσεις που εκφράσατε στα πλαίσια της διεύρυνσης. Κρατήσατε ζωντανή τη διαδικασία, πιστέψατε στο κεντρικό χαρακτήρα, στον κομβικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και ε, επιμείνατε έτσι ώστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Τούρκους σε βασικούς τομείς. Καταφέρατε να κρατήσετε ζωντανή επίσης και την τουρκική προσπάθεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος Χάν θα συνεχίσει την εξαιρετική σας προσπάθεια και θα συνεργαστούμε εξίσου στενά μαζί του. Όπως είπε η κυρία Μοντγκερίνη, ε, ο δρόμος που ακολουθήσαμε είναι ο καλύτερος, γιατί μακροπρόθεσμα μπορεί να υπάρξουν οι αλλαγές που απαιτούνται σε επίπεδο δημοκρατίας, κράτους δικαίου και οικονομικής ανάπτυξης. Βέβαια, οι ενδείξεις λέγουν ότι υπάρχουν πολλά που να γίνουν στην Τουρκία, ιδιαίτερα σε επίπεδο κράτους δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαχωρισμού της εξουσίας και ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Αυτά είναι και τα θέματα που ενδιαφέρουν τις διαπραγματεύσεις. Τα βασικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις στα κεφάλαια 23 και 24 όπως και εσείς και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα θέλαμε να ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια. Αλλά δεν είναι πιθανό να γίνουν γρήγορα οι βελτιώσεις και διαρωτώ με τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να πείσουμε την Τουρκία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας έκφρασης και στον τομέα του κράτους δικαίου και δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι και εγώ μόλις έχω αναλάβει την ευθύνη για να διαδεχθώ τον προηγούμενο εισηγητή και είναι μια μεγάλη ευθύνη για μένα. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω επί του για μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για την ΑΡΙΜ, για τη ΦΥΡΟΜ και για τις ε, δυνατότητες να συνεχίσουμε την επικοινωνία με τη χώρα αυτή. Θα ακολουθήσουμε τη γραμμή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία περιλαμβάνεται και στην σημερινή σας έκθεση. Είναι σαφές ότι το μείζον πρόβλημα για τη ΦΥΡΟΜ και θα χρησιμοποιήσω αυτό το επίσημο όνομα, αν και η χώρα μου αναγνωρίζει τη χώρα αυτή ως Μακεδονία λέει ο ομιλητής, Το τεράστιο πρόβλημα λοιπόν είναι το πρόβλημα του ονόματος. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια πολύ κακή ατμόσφαιρα γύρω από, τις μελλοντικές, ε, από το μελλοντικό ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας αυτής. Έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε με πιο δίκαιο τρόπο και επαναλαμβάνω αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση προόδου να πω δηλαδή ότι λυπάμαι που δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή, γιατί ε, της αξίζει να γίνει αυτό. Και δεν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις λοιπόν. Και γι' αυτό και οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα αυτή δεν ακολουθούν τις κατευθύνσεις τις οποίες θα επιθυμούσαμε για μια χώρα που έχει ευρωπαϊκές τουλάχιστον φιλοδοξίες. Αναφέρομαι εδώ στις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα, στην μεταχείριση του τύπου γενικά και των μέσων ενημέρωσης και γενικότερα τον πολιτικό πολιτισμό ο οποίος επιδεικνύεται στο εσωτερικό του κοινοβουλίου της χώρας. Σε αυτά τα επίπεδα υπάρχουν ε, αρκετά προβλήματα. Επίσης υπάρχουν και προβλήματα σε σχέση με την ιστορία ή την ψευδοϊστορία της χώρας, λέει ο μιλητής. Γενικά πολλά μένει να γίνουν στο μέλλον και τελειώνω, Πρόεδρε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Ναι, ευτυχώ γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσε και η γειτονά σα να πάρει το λόγο μετά. Η Επίτροπε. Νομίζω ότι όταν ε, κάποιοι συνάδελφοι και ακόμη και ο πρόεδρος Μπαρόζο προσπάθησαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες ε, ήταν ε, κάποια, ότι δείξαμε κάποια σκληρότημα. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώ όταν ήμασταν σκληροί και αυστηροί τότε ήταν που τους υποστηρίζαμε και τους βοηθούσαμε περισσότερο. Και το θέμα δεν είναι μόνο να καταπολεμήσουμε την κόπωση από τη διεύρυνση, αλλά και ένα άλλο φαινόμενο που υπάρχει και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Την κόπωση των μεταρρυθμίσεων, που είναι εξίσου σημαντική. Προσπαθήσαμε να είμαστε δημιουργικοί, ευρηματικοί και να δημιουργήσουμε με συγκεκριμένη δομή και ένα διαρθρωμένο διάλογο για να κρατήσουμε τη φλόγα το, της διεύρυνσης ζωντανή και νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που θα ήθελα να διαβιβάσω προς το διάδοχό μου είναι όχι μόνο να αξιοποιήσει στο έπακρο τους ε, μηχανισμούς που υπάρχουν, αλλά να ε, τους παρουσιάσει και καλύτερα ε, στην περιοχή και να δώσει το παρόν εκεί, δίνοντας έμφαση στην αρρωγή προς τις υποψήφιες χώρες. Είναι εύκολο να λέμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική και μετά να αφήνουμε τις επιμέρους χώρες ή ε, ολόκληρη την περιοχή σε, στη μοίρα τους και να τις αφήνουμε μόνες τους να παρουσιάζουν έργο. Γιατί ο κόσμος θέλει αλλαγέ όχι μετά από 5 και 10 χρόνια, αλλά σήμερα, αύριο, θέλουν από τώρα να δουν τη διαφορά. Και θα πρέπει η δυσκολία και τα δεινά των μεταρρυθμίσεων να αντισταθμιστούν με ορατά και αυτά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επόμενη περίοδο. Και ευελπιστώ ότι το μήνυμα θα το λάβουν οι αρμόδιες αρχές και δεν θα χαλαρώσουν τη δέσμευσή τους, όχι μόνο υπέρ των μεταρρυθμίσεων, αλλά και στην διατήρηση του εσωτερικού διαλόγου ζωντανού. Μία διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς. Και όσο περισσότερο το συζητάμε, τόσο πιο δύσκολο το βλέπουμε στην πράξη. Γιατί παρόλο που ο συμβιβασμό δεν έχει καλή φήμη πολλέ φορέ σε αυτή την περιοχή, σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Γι' αυτό και στην τελευταία έκθεση ήθελα να τονίσω ακριβώ την ευθύνη που φέρουν και οι κυβερνώντε αλλά και η αντιπολίτευση να διαφυλάξουν και να κρατήσουν ζωντανό τον πολιτικό διάλογο με δημοκρατικούς θεσμούς. Και θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Οι δεν θα πρέπει απλώς να αγκιστρώνονται στα αποτελέσματα των εκλογών και όλα τα άλλα να τα αφήνουν στην αντιπολίτευση. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε στην Τουρκία για να μην ε, να αποστρέψει το βλέμμα της από τις μεταρρυθμίσεις. Το τελευταίο δίμηνο είχαμε τρεις σημαντικές αποστολές ε, για την ε, ε, ποινική δικαιοσύνη, την ελευθερία έκφρασης και την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Είχαμε peer review, αναθεώρηση από ομότιμους και από το καλοκαίρι έχουμε συνεχή διάλογο με τους τουρκους εταίρους μας για το πώς θα εφαρμοστούν ε, οι πολλαπλές συστάσεις ε, που προέκυψαν από τις τρεις αποστολές. Και καταλήξαμε σε συμφωνία, σε κοινή αντίληψη μάλλον με τις τουρκικές αρχές, ως προς το εξής. Από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί η διατύπωση αυτών των συστάσεων, θα αποτελέσουν ε, τη βάση για μια σειρά σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, ακόμη και τη βάση ενός οδικού χάρτη για τις αρχές. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι υποκαθιστούμε με τη διαδικασία αυτή τα κεφάλαια 23 και 24. Απλώς είναι ένας τρόπος για να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα θετικά σημεία, την πρόοδο που έχει σημειωθεί και θεωρώ ότι είναι όχι μόνο προς όφελος της Τουρκίας, αλλά και προς το δικό μας συμφέρον να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Και γι' αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε τα κεφάλαια 23 και 24. Και μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμη. Και στο οποίο έχουμε σημειώσει πρόοδο. Αυτό που χάθηκε ιδιαίτερα στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και στις αρχές της τελευταίας είναι να χάσει το κεντρικό του ρόλο το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Τουρκία. Δικαιοσύνη, συγγνώμη, στην Τουρκία. Και, και θα πρέπει η νέα νομοθεσία να φέρει την Τουρκία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να την απομακρύνει. Και η σύγκληση δεν θα πρέπει να αποτελεί καινό γράμμα για μερικούς γραφειοκράτες στην Τουρκία, αλλά να αποτελέσει μια ουσιαστική πολιτική που θα βρεθεί στο επίκεντρο των κυβερνητικών προσπαθειών στον ενταξιακό δρόμο, στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί με τη νέα κυβέρνηση έχουμε και νέες πολιτικές που βάζουν το Υπουργείο αυτό των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο επίκεντρο. Και θα πρέπει πριν να φτάνουν τα νομοσχέδια στη Βουλή να περνάνε από το Υπουργείο αυτό των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που θα ελέγχει κατά πόσο ευθυγραμμίζεται ε, το προσυζήτηση νομοσχέδιο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και Δέσμευση υπάρχει, θα πρέπει να δούμε όμως και συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Για τη Βοσνία Ζεγοβίνη τώρα. Αυτό που ισχύει εδώ και αρκετό καιρό, ότι σταδιακά έχουμε μία μετάβαση, η εκχώρηση των εξουσιών προς τις αρχές του κοσυφοπεδίου, λέει ο κ. Φίλε. Είναι μία ευπρόσδεκτη διαδικασία, γιατί θα πρέπει το κοσυφοπαίδιο να κάνει κτήμα του την διαδικασία αυτή των μεταρρυθμίσεων στο κράτος δικαίου. Και η εκχώρηση εξουσιών, η μεταφεωρά εξουσιών από τη Γιούλεξ στις αρχές του κοσυφοπαιδίου, σημαίνει ότι το ενταξιακό μέσο διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο και περισσότερο ρόλο. ώστε να ισχύσουν ευρωπαϊκά κριτήρια κατά την εχώρηση αυτή. Έχουμε διαρθρωμένο διάλογο με το Κωσυφοπαίδιο για το κράτος δικαίου και με την ενίσχυση αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου και το προς την Ισλανδία για, με την ενίσχυση λοιπόν αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου θα βοηθήσουμε τις αρχές του Κωσυφοπεδίου να ενισχύσουν και τις εξουσίες του συνταγματικού δικαστηρίου. Και τώρα έρχομαι στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Προσπάθησα να το τονίσω και προηγουμένως ότι από κοινού να απευθύνουμε μια έκκληση προς το λαό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ώστε στις επόμενες εκλογές να ψηφίσουν πολιτικούς που θα τους εξασφαλίσουν καλύτερο μέλλον. Καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Θα πρέπει να έχουμε ενωμένη Βοσνία Ζεγοβίνη που θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία και από ομόνια και νέα φωνή. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή και μετά τις εκλογές και η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσουν όσο μπορούν την Βοσνία και Ζεγοβίνη για να ξεπεράσουν αυτό το διέξοδο και να μην διαψευστούν οι προσδοκίες του βοσνιακού λαού. Και στο παρελθόν είχαμε παρόμοια διέξοδο. Και στη Βοσνία και Ριζεγοβίνη έχουμε κάποιους πολιτικούς που προτιμούν τα κομματικά τους συμφέροντα από το εθνικό συμφέρον. Και οι επικείμενες ευρωεκλογέ θα χτυπήσουν καμπανάκι και μετά τις εκλογές ελπίζω να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατό μια κυβέρνηση για να συνεχίσει την προσπάθεια και να κατασκευάσει μια γέφυρα που θενώνει τον Dayton, τη συμφωνία του Dayton με την φάση διεύρυνσης και ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. κύριο Χάουιτ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά τον Επίτροπο. Ε, άνοιξε πολλά κεφάλαια και προσπάθησε σε όλη την προσπάθεια ακριβώς που έκανε να ανοίξει τις νοοτροπίες, να βοηθήσει ε, και τις αλλαγές που είναι απαραίτητος και το συγχαίρω επίσης που κράτησε και θετικό πρόσημο για την ε, έκθεση της ΦΥΡΟΜ αναφέρομαι στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα αλλά και για τα μποϊκοτάς που σημειώνονται στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και σε άλλου είδους ε, αντίστοιχες καταστάσεις. Διερωτώμε λοιπόν και ερωτώ τον Επίτροπο να σχολιάσει κάπως περισσότερο αυτό που είπε για την αποτυχία της Σέρβιας να ευθυγραμμιστεί στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας και ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε ε, ε, για την Τουρκία, να δούμε για την Τουρκία εάν πράγματι έχει βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα στην καταπολέμηση του ίσης στην Συρία. Θα κατανοήσει ο Επίτροπος ότι εμείς ε, είμαστε υπέρ των μέτρων για την οικονομική σταθερότητα, αλλά θα θέλαμε τα μηνύματα των Βρυξελών να μην ερμηνεύονται πάντα από τους λαούς των περιοχών αυτών σαν μηνύματα λιτότητας και δημοσιονομικής αυστερότητας. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπροκ ε, για την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα. Είστε φίλος της διεύρυνσης, είχε απόλυτα δίκιο ο πρόεδρος Μπροκ και νομίζω ότι χρησιμοποιήσατε μια γλώσσα η οποία λέει πάρα πολλά για μας όλους. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της τελευταίας πενταετίας και ποια είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση. Νομίζω ότι ε, εδώ θα πρέπει πέρα από τις συμβουλές που θα δώσετε στον κύριο Χάν, ε, τουλάχιστον κάποιες από αυτές να τις πείτε και σε μας δημόσια. Βλέπω ότι η κυρία Νάιτσα ήρθε ε, τη στιγμή που έπρεπε. Παρακαλώ 1,5 με 2 λεπτά το πολύ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινώντας εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Επίτροπο για την αφοσίωσή του και την εμπλοκή του υπέρ της διεύρυνσης και υπέρ της, ε, ε, της πολιτικής γειτονίας. Οι καλύτερες ευχές μας θα σας συνοδεύουν κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά των τελευταίων πέντε ετών. Πέραν αυτού τώρα και αν δούμε συνολικά την κατάσταση έτσι όπως την περιγράφεται. Βλέπω και μου κάνει εντύπωση ότι πολλές παλαιές διαφορές δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Το είπατε και εσείς, αναφερθήκατε στο θέμα του ονόματος γύρω από τη ΦΥΡΟΜ. Είναι ένα πρώτο πρόβλημα στο οποίο μπορώ να αναφερθώ. Η έλλειψη ενός νέου συνταγματικού χάρτη στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τα προβλήματα ανάμεσα στην Τουρκία και την Κύπρο και υπάρχει βέβαια η καλή εξαίρεση της βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο. Αν δούμε την κατάσταση αυτή συνολικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές οι οποίες φαίνονται παγιωμένες και δεν φαίνεται να αλλάζουν. Διαρωτώ με λοιπόν, κάποια πράγματα θα προτιμούσατε να τα κάνετε με διαφορετικό τρόπο και τι σύμβουλες θα δώσετε στον διάδοχό σας έτσι ώστε τα πράγματα επιτέλους να αλλάξουν και να βελτιωθούν έτσι ώστε να επιληθούν κάποιες από, τις, από τα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Νάιτς Καστάλτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την τεράστια προσπάθειά του και θα ήθελα να ευχηθώ και σε αυτόν και στον επόμενο επίτροπο ότι καλό. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την Τουρκία. Αναφερθήκατε εσείς στη σημασία του κράτους δικαίου στα πλαίσια της διαδικασίας διεύρυνσης. Αναφερθήκατε στις προσπάθειες που έχουν γίνει για μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σώμα που δεν επέτρεψαν όμως να υπάρξει πρόοδος για τα κεφάλαια 23 και 24. Το πρόβλημα για τη χώρα αυτή ίσως να είναι και η έλλειψη της, του ορισμού της έννοιας της τρομοκρατίας και στον παλαιό κώδικα και στον κώδικα του, του 1991 είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και στον ποινικό κώδικα και με τρόπο αντιφατικό σύμφωνα με την Amnesty International αυτή η σύγχυση πολλές φορές χρησιμοποιείται ε, και από τους πολιτικούς για να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον και για να καταδικάζουν μερικές φορές ε, οι δικαστές την απλή συμμετοχή ε, σε κάποιες πολιτικές οργανώσεις, ανεξαρτήτως της χρήση βίας ή όχι. Το θέμα λοιπόν κάποιων αλλαγών και για το καθεστώς των κομμάτων έχει παγώσει στο Κοινοβούλιο, δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Και επίσης υπάρχουν και επανειλημμένα ακούγονται απειλές εις βάρος των κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι γίνεται με τον οδικό χάρτη στον οποίο αναφερθήκατε λίγο, τι προοπτικές υπάρχουν στα πλαίσια της νοοτροπίας more for more, έτσι ώστε να αλλάξει με θετικό τρόπο η Τουρκία και να κάνει επιτέλους τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Φιούλε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την δέσμευση και την αφοσίωση σας στη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε 11 πριν, τώρα 12 ε, Κροάτες Ευρωβουλευτές που αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας σας ε, στο χαρτοφυλάκιο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν σε μια προβολή μια της επιστολής για, συνεργασία, για τις εργασίες στον, στον Επίτροπο Χάνα να μου πείτε τι θα τον συμβουλεύατε για να συνεχιστεί αυτή η πορεία επιτυχίας, success story και επίσης να μου πείτε τι περιμένετε μετά τις εκλογές στη Βοσνία Ριζεγοβίνη και τη θέση των Κροατών ως την πιο ολιγάριθμη αλλά και ευάλωτη ομάδα της χώρας. Για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μιλάω. Τι περιμένετε λοιπόν από τις εκλογές 12 Οκτωβρίου και σταγματικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της θέσεως των Κροατών ως την πλέον ευάριθμη αλλά και ευάλωτη ομάδα, εθνοτική ομάδα της χώρας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, οι διερμηνείς είναι εδώ μέχρι τις δύο μόνο. Οπότε ε, θα περιορίσω τις παρεμβάσεις σε ένα μόνο λεπτό. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη δουλειά του. Πρόσφατα διορίστηκα, ανέλαβα εισηγητής για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Σκιώδησε γιατί συγγνώμη. Ερωτώ λοιπόν ε, αν υπάρχουν προοπτικές μέσα από μια νέα συμφωνία για την χώρα, μια νέα συμφωνία που θα μπορούσε να δοθεί και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω για την πρόοδο που σημειώνεται και εσείς στις χώρες της περιοχής. πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων ώστε να αναλάβουν ε, τις ε, δραστηριότητες, τα καθήκοντα και τις πρωτοβουλίες τους όλοι οι παράγοντες. Τι μπορείτε να προβλέψετε για την σταγματική μεταρρύθμιση, εάν πιστεύετε ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων τεχνοκρατών στη χώρα θα μπορούσε να βοηθήσει με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης μιλήσατε για τα Βαλκάνια, αλλά οι Βόσνοι πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρε πριν από μερικού μήνε ενημερώθηκαν ότι δεν πρόκειται το ΕΠΑ 2 να τους δώσει χρηματοδότηση. Πώς λοιπόν θα εξασφαλιστεί αυτή η υποστήριξη. Ευχαριστώ. E Ω συντονιστή των συντηρητικών μεταρρυθμιστών μιλάω λέει ο κύριος Κινοκνεύ ναι, και εγώ συμφωνώ για το θέμα της ονομασίας, ε, το σταγματικό αδιέξοδο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα ήθελα να αναφερθώ ωστόσο στην Σερβία μαζί με την Τουρκία που δεν υποστηρίζει τις ε, κυρώσεις κατά της Ρωσίας αλλά και που ε, ακολουθεί το, μια στάση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως προς την αναγνώριση της Ε, Κρυμαίας, της αυτονομίας Κρυμαίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι για την ε, Τουρκία τώρα που υποχρεούται η, η Κύπρος λόγω των αναπτυσσόμενων ερευνών για υδρογονάνθρακες στα ανοιχτά της Κύπρου και επιχρόνοντας εκ τούτου οι Κύπροι να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι έχετε να πείτε για την ε, σχέση τους με την ΆΕΣΙΣ και τι έχετε να πείτε για την Αρμενία. όρος... Στα πλαίσια λοιπόν της Επιτροπής Μπαρός, ο όρος αυτός ήταν πολιτικά ορθός. Αναφερθήκατε επίσης στις δυνατότητες που έχει η διεύρυνση να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε κάποιες χώρες δεν υπάρχουν πολλά κίνητρα για μεταρρυθμίσεις. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες νέες δυνατότητες προς την κατεύθυνση αυτή μπορείτε να δώσετε στις χώρες αυτές νέα μέσα και νέες μορφές οικονομικής στήριξης έτσι ώστε να νιώσουν οι χώρες αυτές ε, κάποια κίνητρα, κάποια βοήθεια. Και τέλος, μια περίεργη παρατήρηση ίσως. Ένα περίεργο πράγμα. Ε, ε, όλοι οι επίτροποι για τη διεύρυνση έχουν τέσσερα γράμματα στο επίθετό τους και οι τρεις τελευταίοι. Είναι μια ιστορική σύμπτωση και ελπίζω να βοηθήσει τον κύριο Χάν να ακολουθήσει τις σωστές πολιτικές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φιούλερ για την ενημέρωση και εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε. Όπω εσεί ο ίδιο επισημαίνετε, έχει υπάρξει σαφή οπισθοδρόμηση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία σε κέριου τομεί όπω του κράτου δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, των μέσων μαζική ενημέρωση, τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και ούτω καθεξή, και άρα δεν πληρούνται τα κριτήρια τη Κοπεχάγη κατά το τελευταίο έτο. Για να μην αναφερθώ σε ακραίε εθνικιστικέ και επεκτατικέ θέσει που εκφράζονται από επίσημα κυβερνητικά χείλη, οι οποίε σε καμία περίπτωση δεν προάγουν τι σχέσει καλή γειτονία. Εν τούτη τη σύστασή σα προς το Συμβούλιο προβαίνεται σε ένα θεσμικό ακροβατισμό θα έλεγα, προτείνοντας την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων επί τη βάση τη αθρηστική προόδου τη χώρα κατά τα τελευταία έτη. Πείτε μου σα παρακαλώ, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η επιβράβευση τη κακυποψήφια χώρα, δεν αποτελεί αυτό αντιστροφή της αρχής της αιρεσιμότητας που είναι ο ακρογωνιαίος λήθο της διαδικασίας διεύρυνσης δεν υπάρχει κίνδυνος αυτό να αποτελέσει κακό προηγούμενο και για άλλες χώρες που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ehm, godātais komisār kungs, es īsti negribētu piekrist, kad piecu jūsu gadu. Ευχαριστώ. Desinfono. Oti. ότι η πενταετή θητεία σας ήταν μια success story, ήταν μια πολύ πετυχημένη. Σίγουρα η ένταξη της πελατείας ήταν σημαντική επιτυχία, αλλά έχω συνομιλήσει με ε, σημαντικούς αξιωματούχους της Τουρκίας που μου είπαν ότι ένας από τους λόγους που αποστασιοποιείται και απομακρύνεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το γεγονός ότι η η Ευρωπαϊκή Ένωση ταπεινώνει την Τουρκία με τον τρόπο που χειρίζεται τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Στη διάρκεια της θητείας σας, ε, κύριε φίλε, ε, τα σύνορά μας με το Αζερβαϊτζάν ε, βρέθηκαν σε κίνδυνο και το Αζερβαϊτζάν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν λοιπόν όλα ρόδινα στην θητεία σας έχουμε αρκετέ ε, μορφέ να σα προσάψουμε και ίσω και έναν οδικό χάρτη θα μπορούσαμε στην περίπτωση αυτή. Την ερώτηση δεν την κατάλαβα. Τι περιμένετε από μένα. Δεν ήταν ερώτηση, ένα σχόλιο ήταν απλώς. Ε, Ο κύριος Έμπερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Εγώ πιστεύω ότι για να ολοκληρώσουμε τη διεύρυνση προς Ανατολάς θα πρέπει να τη θέσουμε ως την προτεραιότητα γιατί έχει μεγάλη σημασία και από πολιτική και από οικονομική άποψη. Βέβαια η ένταξη είναι προτεραιότητα για πολλές χώρες και δεν έχουμε εντυπωσιακή πρόοδο σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχει μια συμμετρία και μια διαφορά στην πρόοδο των διαφόρων υποψηφίων χωρών. Θα πρέπει να προωθήσουμε το στρατηγικό μας πρόγραμμα σε όλη την περιοχή, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επιμέρους ευαισθησίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και επίσης θα πρέπει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις σε εκρεμή και ανεπίλητα διμερή ζητήματα. Και σίγουρα να ενθαρρύνουμε τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν μεταξύ τους. Πιστεύετε ότι με μια ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας θα έχουμε μια πιο ομοιόμορφη πρόοδο στην ενταξιακή πορεία των χώρων αυτών και ποιες είναι οι προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Κύριε Φούλε, η αρχική σας δήλωση What is the advantage of the hearings? Ξέρετε ποιο είναι το πλεονέκτημα των ακροάσεων? Είναι ότι δεν χρειάζεται ο υποψήφιος επίτροπος να σημειώνει α, τις ερωτήσεις στο χαρτί. Ξέρω ότι είστε εδώ σε έχετε, έχετε μπει σε ρυθμού ακρόαση, αλλά θέλω λίγο χρόνο για να μπορέσω να προλάβω να σημειώσω τις ερωτήσεις και να τις απαντήσω. Με πιέζει βέβαια με το χρονόμετρο συνέχεια ο Έλμαρ. Αν θέλετε να απαντήσω, αφήστε μου χρόνο να σημειώσω τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε σε ένα λεπτό να υποβάλουμε ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο. Ο Τσάρλ είναι αστέρι στην ταχύτατη υποβολή ερωτήσεων. Να επικεντρωθείτε. Μία-δύο ερωτήσεις το πολύ. One minute. Καλώς, να κρατήσω λοιπόν αυτό τον κανόνα του ενός λεπτού. Η πολιτική διεύρυνση δεν είναι ένα κούτι της Πανδώρας. Όπως είπατε και στην ομιλία σας σήμερα, υπάρχουν ορισμένες, ορισμένοι κανόνες. Οι κοινοτικοί κανόνες καταρχάς. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Βλέποντας τις τελευταίες ε, εξελίξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου με, τις στρατιωτικές, ε, με το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας το οποίο παρεμβαίνει και παρεμποδίζει ε, την Κυπριακή Δημοκρατία να αναζητήσει φυσικό αέριο. Πιστεύετε πράγματι ότι μια υποψήφια χώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία, σέβεται το κοινοτικό δίκαιο και τους βασικούς θεμελιώδεις κανόνες. Και δεύτερον, ε, εσείς αν πρέπει να προτιμήσετε θα ε, υπερασπιστείτε κάποιες άλλες πολιτικές ή το κράτος δικαίου όπως το πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη ερώτηση για το κοσυφοπαίδιο. Για να γίνει μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απαιτείται ομοφωνία. Γνωρίζετε ότι η Ισπανία δεν αναγνώρισε το κοσυφοπαίδιο. Οπότε τι νόημα έχει η έναρξη συζητήσεων αν μία από τις χώρες μέλη, εν προκειμένου η Ισπανία, δεν αναγνωρίζει την υποψήφια για ένταξη χώρα. Δεύτερον, θεωρείτε, πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν συμφέρον να, ε, να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης πιστεύετε ότι η Τουρκία ε, οι Τούρκοι πιστεύουν ότι από τη στιγμή που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και φαίνεται ότι η εταξιακή πορεία της Τουρκίας μοιάζει με την διαδικασία του Όσλο, δηλαδή δεν οδηγεί πουθενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Φούλε. Είχαμε πολλές συναντήσεις, πολλές διαφωνίες κατά καιρού, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ τη συμπεριφορά, την ευθύτητά του πάνω στα ζητήματα που συζητούσαμε. Ε, την πρώτη μου ερώτηση την έχει καλύψει ο κύριος Τάνο και ο κύριος Μαυρίδης, δεν θα την επαναλάβω, μια γραμμή μόνο. Δεν σχολιάσατε καθόλου την επέμβαση της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου με αποτέλεσμα την διακοπή των συνομιλιών. Το δεύτερο που έχω να πω, κατά την κρίση μου, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοροϊδεύουν την Κύπρο όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού και άλλες κοροϊδεύουν την Τουρκία. Εσείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσατε σαν θεσμοί να βρείτε έναν τρόπο να μπείτε πάνω σε αυτό το ζήτημα γιατί συζητάτε και το άνοιγμα των κεφαλαίων 23-24 χωρίς να τα διασυνδέετε καθόλου με το κύριο γεγονός που δεν επιτρέπει το άνοιγμα τους που είναι το κυπριακό είτε εσείς είτε η κυρία Πύρη. το να αποφεύγει να δει κανείς την πραγματικότητα δεν την επιλύει. Θέλω λοιπόν να ξέρω μπορούσατε να κάνετε κάτι παραπάνω ή όχι. Ο David Cameron, κύριε Επίτροπε, μιλάει για μια Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ατλαντικό στα Ουράλια αλλά με, την, ε, με τις επιδόσεις ε, μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπω καμιά σπουδαία πιθανότητα να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο και βλέπουμε μια τεράστια μετανάστευση η οποία μειώνει το γενικό ΑΕΠ κατά κεφαλή, μια τέτοια πολιτική η οποία δεν εντάσσεται στις προοπτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ τη ελεύθερη διακίνηση και ελπίζω ότι θα μπορέσει ο διαδοχό σα να διευκρινίσει κάποιε από τι τοποθετήσει του, προκα... Ε, του δικές σας για την επέκταση όλο και περισσότερο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτό αυτό ανεξαρτήτως συνεπειών. Βεβαίως χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και το οικονομικό και το δημοκρατικό βάρος και άθο που επιβαρύνει τη χώρα μου ως προς τα προβλήματα που δημιουργεί για την ευημερία η όλο και μεγαλύτερη διεύρυνση και προφανώς αυτό δεν βοηθάει στο να καταστεί πιο δημοφιλής Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστώ τον Επίτροπο Φιούλε για τη δουλειά του τελευταία αυτά πέντε χρόνια. Ε, και εδώ αλλά και στα Βαλκάνια, στις, στα Δυτικά Βαλκάνια έχει τύχει ιδιαίτερη αναγνώριση αυτή η στάση του. Έχει συμβάλει κατά τρόπον αυτό σε ουσιαστικές εξελίξεις στον τομέα της διεύρυνσης πολιτική του και θα ήθελα ιδιαίτερως να υπογρομίσω τρεις ανησυχητικές εξελίξεις που επεκτείνονται στην περιοχή και που με ανησυχούν. Ο ρόλος, η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και ο πολιτικός διάλογος. Εδώ λοιπόν χρειάζεται περισσότερο δραστήριο ρόλος από πλευρά μας, από τα μέλη δηλαδή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διευκολύνουμε τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των εταίρων μας στην περιοχή, αλλά χρειάζεται συντονισμό συνεργασία μεταξύ των πολιτικών πολιτικών ομάδων σε αυτό το κοινοβούλιο για να αποστείλουμε μηνύματα που θα είναι τα ίδια με την ίδια διατύπωση και αυτό το λέω προς άπαντα ακούοντα. Επίσης, το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και βέβαια τρίτον η ε, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά. Η οικονομική διακυβέρνηση έχει μεγάλη σημασία και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, χαίρετε κύριε Επίτροπε, αντίο και ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ε, επιτυχημένη θητεία σας και ε, να σας ευχαριστώ όχι μόνο για την πατρίδα μου που σήμερα γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας αλλά ε, να σας ευχαριστήσω και για των γειτονικών χωρών. Είναι δύσκολη η κατάσταση για τη διεύρυνση, έχουμε πολλές προκλήσεις αλλά δεν θεωρώ όμως ότι η εμβάθυνση και η διεύρυνση είναι ε, αντίπαλες διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι ε, η διεύρυνση θα πρέπει να προωθηθεί μέσω της ασφάλειας, της συνεργασίας και ε, αντίληψη καλύτερα της κατάστασης ε, και στα σύνορά μας. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν θα πρέπει μόνο να σταθεροποιήσουμε την πολιτική γειτονία μας, αλλά να σταθεροποιήσουν και οι γείτονές μας τη δική τους κατάσταση. Θεωρείτε ότι οι απειλές ως προς την ασφάλεια εξαιτία της σύγκρουσης στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και στη Μέση Ανατολή θα επιβαρύνουν τη διαδικασία της διεύρυνσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για Τουρκία υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. 15 χρόνια τώρα ασχολούμαι με τη χώρα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν από το 1999 μέχρι τώρα κάποιε μεταρρυθμίσει, αλλά ε, χάθηκαν πολύ γρήγορα μετά το 2005 και την αναγνώριση του κράτους ε, ω την έναρξη των διαπραγματεύσεων καλύτερα. Ιδιαίτερα οι τελευταίες τρει ε, εκθέσεις προόδου καταγράφουν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σαφέστατα αυτή την επιβράδυνση. Νομίζω ότι η Τουρκία δεν μας παίρνει καθόλου στα σαβαρά, δεν θέλει να προσχωρήσει με τους όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να προσχωρήσει σαν να κάνει το χατήρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το υπερβάλλει λίγο. Η Τουρκία νομίζω ότι έχει ορίσει τους δικούς τους κανόνες. Δηλαδή λέει θέλουμε να μείνουμε όπως είμαστε και έχουμε τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση που εσείς όπως και να έχει κάποια στιγμή θα μα αποδεχθείτε όπως είμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να αλλάξει και όχι η Τουρκία δηλαδή. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί εμένα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να είναι όλο και πιο διατεθειμένη να ξεπουλήσει την ευρωπαϊκή της ψυχή, το ευρωπαϊκό της πνεύμα, τις αξίες για να κερδίσει το στρατηγικό εταίρο την Τουρκία με μια προοπτική ε, διεύρυνσης, δηλαδή. Τι γνώμη έχετε σε αυτά. Μογκερίνη την προηγούμενη Δευτέρα κατά τη διάρκεια των ακροάσεων είπε ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηρίζονται στους κανόνες δικαίου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η στάση απέναντι στην Τουρκία δεν αποδεικνύει αυτή την τοποθέτηση της κυρία Μογκερενή και αντίθετα βλέπουμε αντί να προσπαθεί η Τουρκία να προσαρμοστεί στις αρχές και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στις αναχρονιστικές και επεκτατικές πολιτικές της ίδιας της Τουρκίας. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Φούλε, και εγώ σας ευχαριστώ για τα πέντε χρόνια που συνομιλούσαμε. Βεβαίως, πάντα μου δίνατε την ίδια στερεότυπη απάντηση. Όταν θα λυθεί το Κυπριακό, όλα θα διορθωθούν. Ελπίζω σήμερα να είναι διαφορετική η απάντηση σας. Είναι η τελευταία ερώτηση που σας υποβάλλω. Δεν αναφέρεται λέξη για την δήλωση Τσαβούσογλου, η οποία κατατέθηκε στις 23 Ιουνίου στο ε, Συμβούλιο Σύνδεσης για με την κατηγορηματική θέση της Τουρκίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει, έχει εκλείψει, is defunct. Θέλω να τοποθετηθείτε για αυτό το ζήτημα, αν μπορεί αυτό να συνάδει με την συμπεριφορά ενός κράτους δικαίου και περιμένω την απάντηση σας στο ερώτημα του κυρίου Μαυρίδη. Δηλαδή μπορεί να στέλνει το στόλο γύρω από την Κύπρο και να θεωρείτε ότι αυτό είναι δημοκρατία, είναι κράτος που μπορεί να ε, ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια μικρή ερώτηση. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Λέω πρόεδρος χωρίς το μικρόφωνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς τα δημοκρατικά δικαιώματα της ε, κοινοβουλευτικής μειοψηφίας στην Αλβανία. Προβλήματα που συνεχίζονται. Και σημαίνει ότι δεν έχουν δικαιώματα στην πράξη οι θεσμοί αυτοί, αλλά και άλλοι θεσμοί. Αλλάζει το προσωπικό ε, στις υπηρεσίες φανταζόμαστε ότι εννοεί ο μιλητή με κάθε αλλαγή κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Δεν πληρούνται λοιπόν οι όροι του κράτους δικαίου. Αυτό τώρα που σας εξέθεσα ως ε, διαπίστωση αληθεύει ή όχι. Ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Uh, uh, για να ξεκινήσω με την Αλβανία. Ε, έκανα την παρατήρησή μου κατά τρόπο πιο γενικό, αλλά κατά τον τελευταίο διάλογο και τις συστήσεις που είχα στα Τύρανα, κατέστησα απολύτως σαφές ότι η απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου για το θέμα αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Και δεύτερον, και είναι αυτή η προτεραιότητα, πρέπει να έχουμε δηλαδή την υποχρέωση, ότι έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέπουν στην αντιπολίτευση να ασκεί τα δημοκρατικά της δικαιώματα. Συζητήσεις έχουν γίνει για την ανεξαρτησία και άλλων θεσμών στη χώρα. Η θέση μου είναι ότι όποιε αλλαγέ και να προχωρήσουν θα πρέπει οι θεσμοί αυτοί να παραμείνουν διαφανεί, να λειτουργούν με σεβασμό στο κράτο δικαίου και την νομοθεσία. Και έχουμε, όπως ξέρετε, μία μακροπρόθεσμο χαρακτήρα αποστολή προσωπικού στην ε, Αλβανία με επαφές στην ε, ε, χώρα με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Πάνε και έρχονται συνεχώς και προσχωρούμε και στην οργάνωση σεμιναρίων ώστε να υπάρξει σχετική ενημέρωση και βέβαια ανάλογα θα διατυπώνω και εγώ τις συστάσεις μου εδώ. Κοιτάξτε, είτε είμαι εδώ, είτε μιλάω με την πλειοψηφία, είτε μιλάω με την μειοψηφία στην Αλβανία, είτε μιλάω με τις μειονότητες, είτε μιλάω με την ευρύτερη κοινωνία, οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα και να κάνω είναι σημαντικό για την διαδικασία. Η διαδικασία της διεύρυνσης δεν στηρίζεται μόνο σε μία μονομερή προσέγγιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους λέμε ότι θέλουμε με τις συζητήσεις αυτές να έχουμε μια ως δυνατόν ευρύτερη εικόνα και άνοιγμα της χώρας και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και αλληλεπίδραση με όλους τους φορείς. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει βιώσιμη πρόοδος χωρίς ιδιαιτέρως η πλειοψηφία και η μειοψηφία της ε, Βουλής να συμφωνήσουν σε μια ευρωπαϊκή ατζέντα, σε ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο που θα αποτελεί για αυτούς μια πλατφόρμα όχι μόνο για ανοιχτή αλλά και για συνενετική προσέγγιση. Εγώ έχω δεσμευτεί να καταπολεμήσω την ιδέα αυτή ότι ε, οι εκλογές είναι το άπαν και άπαξ και γίνουν οι εκλογές και εξασφαλίσει το κόμμα την πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του χωρίς καμιά αντίδραση. Όχι, γιατί υπάρχει μειοψηφία, υπάρχει αντιπολίτευση και πρέπει και αυτής η άποψη να λαμβάνεται υπόψη και πρέπει να δημιουργούνται οι σχέσεις εκείνες, οι βάσεις εκείνες για να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Αυτό όχι μόνο γιατί μπορεί να χάσει το ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές την εξουσία, αλλά γιατί οτιδήποτε κάνει στην υλοποίηση της εντολής που θα του δώσει ο λαός δεν θα μπορεί να διατηρηθεί εάν δεν έχει στηριχθεί σε μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία. Είχαμε και διάφορες ερωτήσεις για την Κύπρο καταρχήν και τις ε, τουρκικές δραστηριότητες κάποια γεγονότα, κάποιες δηλώσεις και μια ρηλουχία γεγονότων που οδήγησαν στην απόφαση ε, να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση. Μίλησα για την κατάσταση αυτή στην εισαγωγική μου ομιλία. Το μόνο που έχω να προσθέσω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να διαβάσουμε την έκθεση πρόοδου που επαναλαμβάνει την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα κυρίαρχα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, επιμέρους χωρών να έχουν συμφωνίες για τις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες και να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους ε, και τον πλούτο τους που βρίσκονται στα χωρικά τους ύδατα και στα εδάφη υπό την... που εμπίπτουν στην κυριαρχία τους και με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο. Αυτό που λέει η έκθεση πρόοδου και το επανέλαβα και εγώ στην αρχική μου ομιλία είναι ότι υπάρχει ανάγκη για μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος. Αυτό το είπα και στην αρχή. Πάντως, ε, όταν μαζί με τους συναδέλφους ε, πριν από μια πενταετία έθεσε το ζήτημα της αξιοπιστίας, δεν θέλω να πω ότι η αξιοπιστία τους δεν στηρίχθηκε σε μια γραφειοκρατική διαδικασία όπου εμείς προσπαθήσαμε να ξεγελάσουμε την, τις υποψήφιες χώρες ή να ξεγελάσουμε τα κράτη-μέλη, να τους κοροδέψουμε. Νομίζω ότι δήλωσα σαφώς και κατηγορηματικά ότι η διαδικασία διεύρυνση θα ανακτήσει την αξιοπιστία της όταν ξαναθέσουμε στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής τις θεμελιώδεις μας αξίες και αρχές. Γιατί σε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στο κράτος δικαίου, την λογοδοσία, την ανεξαρτησία της, της δικαιοσύνης, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και τα έφερα στο επίκεντρο και της δικής μου προσπάθειας. Γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικές καμπές. Καταρχήν, πετύχαμε η διαδικασία διεύρυνση να μην είναι μια τυπική διαδικασία που απλώς θα συμπληρώναμε ε, μερικά κουτάκια ότι αυτό το κάναμε, αυτό το κάναμε. Δεν αρκεί μια τέτοια διαδικασία. Βλέπουμε τις επιδόσεις και εξακριβώνουμε κατά πόσο εφαρμόστηκε η νομοθεσία και κατά πόσο οι θεσμοί είναι ανεξάρτητοι από πολιτικές επιρροές. Αυτό λένε τα κεφάλαια 23 και 24. Γιατί οι χώρες που έχουν ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις, σε αυτό το θέμα θα πρέπει να επικεντρωθούν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Αυτά τα κεφάλαια. Και δεν είναι μόνο η μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου μιας χώρας που μας ενδιαφέρει, αλλά και η αλλαγή στην οτροπία. Και αν με ρωτήσετε ποια είναι από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα, ποτέ δεν ξέχασα για ποιον εργάζομαι. Εγώ υπηρετώ τα κράτη-μέλη. Εσάς υπηρετώ. Για σας δουλεύω. Μου αναθέσατε όμως μία εντολή. Να μη φυσώ προσπαθειών προκειμένου η διαδικασία διεύρυνση να μην γίνει ει βάρο των αρχών και αξιών μας. Γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό έχει και τόσα σκαμπανεβάσματα. Δεν υπάρχει εδώ αυτόματος πιλότος. Είναι ένα τομέα που κατεξοχήν δεν ε, χωράει αυτόματος πιλότος. Ούτε επέκλειναν ποτέ από αυτά τα ιδεώδη και αυτές τις αρχές και τις αξίες κράτος δικαίου, αρχές και αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά βρέθηκαν από την αρχή και εξακολουθούν να είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσης. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις επίσης για την Τουρκία. Η διαδικασία είναι μια διαδικασία που παραμένει ανοιχτή. Πριν πέντε χρόνια με είχατε ρωτήσει αν ε, μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι η Τουρκία και βλέπω ότι είναι μια διαφορετική Τουρκία και στα πλαίσια μιας διαφορετικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κατανοώ ότι το θέμα δεν είναι μόνο οι αξίες που είναι το πιο σημαντικό βέβαια θέμα, το θέμα είναι να κατανοήσουμε και την, ε, τον μετασχηματισμό της χώρας σε χώρα μέλος κάποια στιγμή αλλά και να κατανοήσουμε το δυναμικό απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσει τις πολιτικές τις οποίες έχει η ίδια χαράξει. Και γι' αυτό ακριβώς Είχα την τύχη κατά τη διάρκεια της εντολής μου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα και στην περίπτωση της Κροατίας και νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε την πολιτική μας και καταλήξαμε στα σωστά συμπεράσματα. Είναι επίσης σαφές ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ε, διεύρυνσης, δεν το κρύβουμε, αλλά πρέπει να είμαστε εδώ ειλικρινείς και θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι όταν υπάρχουν δύο θέματα ανάμεσα σε δύο υποψήφιες χώρες ή σε μία χώρα υποψηφία και σε μία άλλη που θέλει να γίνει υποψήφια, Πράγματι ε, μπορεί να βοηθήσει η διαδικασία ε, διαβούλευσης, η διαδικασία διαπραγμάτευσης, ε, ο διάλογος ανάμεσα στο Κωσυφοπέδιο και τη Σερβία διευκολύνθηκε από την στροφή αυτών των χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν το θέμα αφορά μια υποψήφια χώρα και μια χώρα μέλος, εκεί το θέμα είναι πιο περίπλοκο. Ε, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε τα απαιτούμενα μέσα που χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να αντιμετωπίσει το θέμα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Και επανειλημμένα ζητούμε από τα κράτη-μέλη και από τους αρχηγούς των κρατών μελών να βοηθήσουν έτσι ώστε και οι χώρες μέλη φυσικά να βοηθηθούν και οι υποψήφιες χώρες να ασχοληθούν με θετικό τρόπο με τις εκκρεμότητες, με τα χαίνοντα θέματα. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και τα Ηνωμένα Έθνη. ένα κάτι καινοτόμο στην έκθεση αυτή που σας έχουμε ε, καταθέσει είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το κεφάλαιο 31. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην παρούσα φάση στην Ανατολική Ευρώπη επηρεάζουν βέβαια και εμάς. Είναι σαφές αυτό. Επηρεάζουν και τα Δυτικά Βαλκάνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. δεν μπορεί να υπάρχει μια ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς νόμου σε ένα τμήμα της Ευρώπης και να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει αρνητικά την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας θίγει και εμάς. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι και μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια και νομίζω ότι και η νέα ε, υπεύθυνη ε, θα ακολουθήσει τη γραμμή αυτή, μπορούμε να ανοίξουμε το 31 που ασχολείται με τα θέματα ΚΕΠΑ νωρίτερα στη διαδικασία από ό,τι το κάνουμε τώρα. Και αυτό γιατί. Έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερη διαδραστικότητα ανάμεσα στους, διεθνούς, στους διεθνείς εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Εγώ δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από, ένα, από μια φράση η οποία λέει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η βαθμιαία, η σταδιακή ευθυγράμμιση της τάδε χώρας με τις πολιτικές μας. Είτε αυτό αφορά το σεβασμό κυρώσεων είτε ε, κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι το άνοιγμα του 31 θα μας δώσει την δυνατότητα να ενισχύσουμε τον διάλογο με τις χώρες αυτές και θα επιτρέψει στις υποψήφιες αυτές χώρες ήδη σε μία φάση προημότερη να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να ευθυγραφιστούν με τις δικές μας πολιτικές. Οι κανόνες βέβαια παραμένουν οι ίδιοι η βαθμιαία, η σταδιακή ευθυγράμμιση είναι το αναμενόμενο από πλευράς των εταίρων μας. Εγώ το έχω σημειώσει αυτό επανειλημμένα και στους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Πρέπει να αναστρέψουν την τάση η οποία επικρατεί Δηλαδή αυτή τη στα, την βαθμιαία α, ευθυγράμμιση μερικές φορές τη χρησιμοποιούν αμφίδρομα και αυτό δεν είναι αποδεκτό από μας. Δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε ε, συναποφασίσει για να ξεκινήσει άλλωστε αυτή η διαδικασία. Για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο. Έχουμε επενδύσει πολύ περισσότερη ενέργεια εκεί για την κοινωνία των πολιτών. Εξετάσαμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών τα προβλήματά τους και τη απουσία αποφασιστικότητας της πολιτικής τάξης να προχωρήσει τη χώρα, να κάνει τη χώρα να προχωρήσει, η κοινωνία των πολιτών ενδιαφέρεται για πολλά κοινωνικά θέματα και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Εγώ διεύρυνα άλλωστε τον διαρθρωμένο διάλογο για το δικαστικό σώμα στη Βοσνία Ευζεγοβίνη με συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών και καλύπτοντας και άλλα σημαντικά θέματα του κράτους δικαίου όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς. Και θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και μετά τις εκλογές στην Βοσνία Ευζεγοβίνη. I, uh, Και τελευταίο θέμα η τελευταία ερώτηση που θα απαντήσω, παρόλο που δεν απάντησα σε όλες τις προηγούμενες, και αν θέλετε συγκεκριμένες απαντήσεις, στείλτε μου την ερώτησή σας γραπτός και θα σας απαντήσω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Ε, τι ήταν σημαντικό, τι με ικανοποίησε και τι με δυσαρέστησε. ποτέ δεν ε, περιέγραψα την ε, πολιτική μου με τον όρο της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Μπήκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα όραμα. Το όραμα να κάνω τη διεύρυνση την σημαντικότερη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να φέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες που ανάλαβαν τις ευθύνες από την πρώτη στιγμή και δέχτηκαν τις ε, αποστολές συνεργασίας και ελέγχου. Και χαίρομαι που κατά το πέρυσι της πενταετίας έχουμε μία μεικτή εικόνα. Δεν ε, είμαι ικανοποιημένος, δεν χαίρομαι που μερικοί εταίροι μας χρησιμοποίησαν την ευκαιρία σε μεταρρυθμίσεις και σημειώνουν πρόοδο. Και προβληματίζομαι και ανησυχώ που κάποιες δεσμεύσεις μας έχουν μείνει μετέωρες και με μερικές χώρες βρισκόμαστε σε κατάσταση αδιεξόδου. Τώρα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι περισσότερο. Αυτό θα μου γίνει η ιδέα και αυτό το ερώτημα θα με στοιχειώσει και στο μέλλον. Αλλά αυτό αφού εγκαταλείψω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η τελευταία σου φράση ήταν πολύ σωστή, πολύ εύστοχη και πολύ σημαντική. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Δεν είναι όλα ρόδινα και δεν γίνονται όλα πρόσκοπτα. Αλλά θα πρέπει να εμείνουμε στην προσπάθεια να διατρανώσουμε τις θεμελιώδεις μας αρχές και αξίες, γιατί όπως είπαμε και για την Ουκρανία, το θέμα είναι οι αξίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μας ενδιαφέρει και θα ήταν αδιανόητο να υποαναχωρήσουμε σε σχέση με τις αξίες μας. Θα συνεχίσουμε πάντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την προοπτική κάποια στιγμή οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η επόμενη πενταετία θα είναι μία περίοδος που περιμένουμε πρόοδο και μεταρρυθμίσεις. Και για να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να δούμε και προσπάθειες κριτήρια της ε, Κοπενχάγης και φυσικά τη δυνατότητα απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να εφομοιώσει νέα μέλη. Και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον άρρηκτο τμήμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν στις υποψήφιες χώρες. Αλλά και τα θέματα της διαφθοράς, καταπολέμησης του εγκλήματος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με επαγγελματισμό όλες αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ για την έκθεση, σας ευχαριστούμε για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα τα πούμε ίσως στο Στρασβούργο.